So, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι. τέσσερις και τέσσερα. Καλό είναι να ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Θεμάτων στη νέα μας θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα Να καλωσορίσω και αυτούς οι οποίοι ήταν και στην προηγούμενη θητεία, τα προηγούμενα πέντε χρόνια εδώ πέρα και έκαναν πολύ καλή δουλειά και να καλωσορίσω και όσους ε, εξελίξαν για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο ή είναι για πρώτη φορά τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη τη σημαντικής αυτής επιτροπής. Όταν λέω σημαντική επιτροπή, αυτό σχετίζεται με το ότι η επιτροπή μας κατά την άποψή μου, είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή γιατί ε, εμείς αποφασίζουμε πώς θα διατεθούν πολλά κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και έχουμε ε, άρα δουλειά η οποία πρέπει να γίνει με τρόπο σοβαρό και διακομματικό. Και κατά την εμπειρία μου τα τελευταία πέντε χρόνια η Επιτροπή αυτή εργάζεται με έναν τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει τα σημαντικά ζητήματα της ε, περιφερειακής ανάπτυξης, της ε, συνοχής, της διασυνοριακής ε, συνεργασίας με συμφωνία και συνεργασία. Και αυτή ήταν η δύναμη της Επιτροπής μας. Ακριβώς αυτή η θέληση για συνεργασία ελπίζω να συνεχιστεί και σε αυτήν την θητεία και με τους ε, νέους συναδέλφους. Τώρα λοιπόν περνάμε στην εκλογή του Προέδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 2.13 του κανονισμού περνάμε στην εκλογή του Προέδρου και των τεσσάρων αντιπρόεδρων. Η σειρά θα είναι η εξής. Θα ψηφίσουμε πρώτα για Πρόεδρο της Επιτροπής, και μετά για τους αντιπρόεδρους. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό, λόγω του κανονισμού, θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματα που αντικαθιστούν βουλευτές και θα είναι στην ψηφοφορία για τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Ανδρέα Κοτσολίνο αντικαθίσταται από την κυρία Ελιζαμπέτα Γκολμίνη. Στο ECR ο Βάλτεμαρ Τόμασεύσκη αντικαθίσταται από την κυρία ε, Ιζαμπέλα Ελένα Κλότς. Στην ΚΟΕ η κυρία Μαρτίνα Μίχελς αντικαθίσταται από τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Παπαδημούλη. Εκεί είναι. Άρα δεν σας αντικαθιστά. Ε, λάθος, μου έχουν γράψει εδώ. Και ε, τους μη εγγεγραμμένους η ο κύριος James Glancy αντικαθίσταται από τον κύριο Nathan Gill. Οπότε, περνάμε στην εκλογή Προέδρου. Πριν ε, γίνει αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, χρειάζεται η κάρτα για τις ε, ψηφοφορίες. Όποιος δεν έχει την κάρτα, έχει ακόμα την δυνατότητα πολύ γρήγορα ε, να πάει να την βρει. Είναι στον τρίτο όροφο οι κάρτες εκεί που είναι και οι θηρίδες σας. Εκεί στα δεξιά. Αν έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας, ε, να δούμε εάν έχουμε απαρτία. Η απαρτία είναι 11 βουλευτές, απαρτία έχουμε. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκλογή Προέδρου. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνω πρώτα είναι το εξής, να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια πρόταση για πρόεδρο της Επιτροπής. Ναι. κύριε Κρέλ. Έχουμε ένα πρόβλημα με ένα από τα μηχανήματα της ε, ψηφοφορίας εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ένας τεχνικός. Ε, ή καθίστε δίπλα. Εντάξει. Η Γκουε, παρακαλώ, να μας προτείνει υποψήφιο. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γιουνούς Ομαρτζή για προεδρία της, ε, την προεδρία αυτής της Επιτροπής. Ε, για τους νέους συναδέλφους οφείλω να πω ότι ο κύριος Ομαρτζή ήταν ε, τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και είναι από την ε, νήσο Ρεωνιών και βεβαίως είναι υπέρμαχος ε, της ε, πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ να παρακαλέσω τον κύριο Ομαρζή να συμφωνήσει. Δέχεστε. Βεβαίως, βεβαίως, λέει ο κύριος Ομαρζή είστε τακτικό μέλος διαπιστώνω και διαπιστώνω επίσης πως έχετε υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την δήλωση του κώδικα συμπεριφοράς οπότε είναι η υποψηφιότητά σας εντάξει να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα τώρα θα πρέπει, ε, αν συμφωνείτε, να περάσουμε σε εκλογή διαβοής, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Παρακαλώ λοιπόν να εκλεγεί ο κύριος Ομαζή, πρόεδρος της Επιτροπής μας. Ich möchte dem Kollegen von Herzen Συγχαρητήρια κύριε Ομαζή. Εύχομαι καλή επιτυχία και σας παραδίδω την Προεδρία. Je vote tout d'abord. Λοιπόν, σας συγχαίρω που εκλεγήκατε και σας ευχαριστώ που με επιλέξατε. Που επιλέξατε να είστε σε αυτή την επιτροπή, την θαυμάσια επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης που είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχή. Η οποία στην ουσία είναι η έκφραση της αλληλεγγύης μας που είναι η βάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ, το, το ελπίζω, στη στήριξή σας, στη στήριξη όλων σας. Και σας διαβεβαιώ ότι πάντα θα σας ακούω με προσοχή όλους και όλες σας, γιατί έχουμε σημαντικές ευθύνες ενώπιον μας. Έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, πολλά σημαντικά θέματα, ήδη και κατά την προηγούμενη θητεία με κλίμα καλής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρετίζω την Επιτροπό Κρέτου γι' αυτό, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα προσπαθεί να προωθήσει τις θέσεις του και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στα επόμενα θέματα Πρέπει να πάμε γρήγορα, γιατί στις 4.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε τώρα, εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Αναφέρθηκαν οι αντιπροματικοί, δεν θα τους επαναλάβω. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθούν άλλα τακτικά μέλη. Και, παρακαλώ, τι υποψηφιότητε έχουμε για την πρώτη αντιπροεδρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ τους ε, νέους συναδέλφους στην Επιτροπή μας και όσοι επανεξελέγησαν. Και να συγχαρώ και εσάς κύριε Πρόεδρε αναλαμβάνετε μια σημαντική θέση ευθύνη, ένα σημαντικό αξίωμα. Από πλευρά ε, του ΕΛΚΟ συντονιστή προτείνω τον κύριο Τσίστοφ Χέτμαν για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Νομίζω ότι θα φέρει σε πέρας ε, με πολύ καλό τρόπο τα καθήκοντά του. Ήταν ε, υφυπουργό για θέματα περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα του. Έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια τη σταδιοδρομία του και καλώ του αδέλφου από τι άλλε πολιτικέ ομάδε να τον ψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρο. Άλλε υποψηφιότητε έχουμε. Όχι. Λοιπόν, όπως και προηγουμένω, νομίζω μπορούμε μπορούμε να τον εκλέξουμε διαβοής, εφόσον βέβαια ο συνάδελφος Χέτμαν δέχεται την υποψηφιότητα. Βεβαίω τη δέχομαι. Πολύ ωραία. Ωραία, μπορούμε λοιπόν να τον εκλέξουμε και να τον παρακαλέσω να έρθει εδώ στο Προεδρείο. Le président provisoire. Λοιπόν, μα θύμισε ο ε, προσωρινό πρόεδρο ε, του κανόνε εκλογή των αντιπρόεδρων, ιδιαίτερα το άρθρο 2.13 του κανονισμού. Θυμίζω λοιπόν ότι το Προεδρείο δεν μπορεί αποκλειστικά να αποτελείται από άνδρες ή από γυναίκες και οι αντιπρόεδροι δεν μπορούν να προέρχονται από το αυτό κράτος μέλος. σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε το προσωπικό της Επιτροπής, υφίσταται κίνδυνος σημαντικός να μην σεβαστούμε τελικώς τους κανόνες της διαφορετικότητας του Προεδρείου και επομένως οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να βρουν λύση επ' αυτού και επομένω προτείνω για την εκλογή του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου αντιπροέδρου να προχωρήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν συμφωνείτε, 22 και 23 Ιουλίου θα συναντηθούμε για να συνεχίσουμε καταρχάς με την ε, ψηφοφορία για την ε, τελική συγκρότηση του Προεδρείου που ήδη συγκροτείται από εμένα και τον συνάδελφο Αυτά μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Με συγχωρείτε ιδιαίτερα που θα επιχειρήσω τώρα την πρόταση αυτή που κάνατε εσείς ε, και φυσικά θέλω να σας συγχαρώ και επισήμως από πλευρά ομάδας μου. Ήθελα λοιπόν να πω ότι, ότι θα μπορούσαμε να εκλέξουμε το δεύτερο και τρίτο αντιπρόεδρο, οπωσδήποτε γιατί δεν θα έχουμε συγκροτήσει ολόκληρο το Προεδρείο. Μπορούμε να εκλέξουμε το δεύτερο και το τρίτο αντιπρόεδρο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κάνουμε δύο ψηφοφορίες ακόμη. Δύο ψηφοφοριούλες. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ο συντονιστής παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε συγχαρητήρια. Και εγώ ήθελα αυτό να ζητήσω να συνεχίσουμε Ε, πρόεδρε, νομίζω ότι αν αναβάλουμε σε αυτό το σημείο θα έχουμε καλύτερες πιθανότητες εξέβρεσης υποψηφίων που να σέβονται τους κανόνες. Η ευθύνη της ισορροπίας των φύλων είναι ευθύνη όλων των πολιτικών ομάδων και όχι μόνο του ΕΛΚ βεβαίως και επομένως εγώ υποστηρίζω τη δική σας πρόταση πρόεδρε. Κοιτάξτε, ως ομάδα ID για τέταρτο αντιπρόεδρο είχαμε υποβάλει την κυρία Ντονάτο που αν δεν άλλαξε φίλο από το πρωί εξακολουθεί να είναι γυναίκα. Τώρα, εάν δεν συμφωνείτε με την υποψηφιότητα Ντονάτο επειδή είναι μέλος του ID, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η τέταρτη πρόταση υποψηφιότητα του τετάρτου αντιπρόεδρου δηλαδή, γυναίκα, υφίσταται. Είχαμε υποβάλει αυτή την πρόταση υποψηφιότητα. Τώρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να η αντίρρησή σα να είναι ότι ανήκει στην πολιτική μα ομάδα και όχι κάτι άλλο. Très bien. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, δεν είναι βέβαιο, αλλά αυξημένος κίνδυνος, το Προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες, λέει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις υποψιότητες που έχουν υποβληθεί. Και θα πρέπει το Προεδρείο μας να το εγκρίνει η διάσκεψη των Προεδρείων Και επομένως είναι το σύνολο της σημερινής ψηφοφορία που μπορεί να μην επικυρωθεί. Γνωρίζω τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ο χρόνος ήταν λίγος, περιορισμένος, ώστε να έχουμε λύσεις καλές λύσεις υποψηφιωτήτων και καλή εξέταση του θέματος από πλευράς των ομάδων των πολιτικών. Αλλά επί της διαδικασίας ψηφοφορίας παρακαλώ να μην επιβαρύνουμε με αυξημένο κίνδυνο διότι διατρέχουμε πράγματι τον κίνδυνο να έχουμε τελικώς τη συγκρότηση ενός προεδρίου που δεν θα σέβεται τους κανόνες για να υπάρξει καλή μελλοντική συνεργασία την επόμενη πενταετία, αποσύρω το έτοιμά μου και ακολουθώ την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντσε. Ε, όντως αναγνωρίζω τον, ε, τη σωστή σας συμπεριφορά. Με τέτοιο πνεύμα θα μπορέσουμε να βρούμε πολύ γρήγορα μία λύση. Για άλλη μια φορά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο και κατόπιν θα κλείσω τις συνεδρίες. Πρόεδρε, εγώ ζητώ εκ νέου να ψηφίσουμε τον τρίτο και τέταρτο υποψήφιο για τους αντιπροέδρους. Επαναλαμβάνω, υπάρχει υποψηφιότητα γυναίκας, υπάρχει υποψηφιότητα γυναίκας. Εκλέξαμε διαβοής τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία και για τον τρίτο και τέταρτο. Je pense avoir été euh, assez euh, explicite. Νομίζω ότι υπήρξα σαφής και ρητός, λέει ο Πρόεδρος. Διακόπτουμε εδώ και θα τα ξαναπούμε 22 και 23 Ιουλίου. Ευχαριστώ όλους.